Dear President, Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα πρακτικά της χτεσινής συνεδρίασης, όπως και τα κείμενα που εγκρίθηκαν, είναι στην διάθεσή σας. Έχετε κάποια αντίρρηση. Όχι. Οπότε εγκρίνονται τα πρακτικά. Πριν περάσουμε στην συζήτηση